τις εργασίες τους εδώ. Οι αρχές της Γαλλίας με ενημέρωσαν για την εκλογή των εξής κυρίων, κυρίων και κυρίων από 16 Μαΐου 2012, Ερίκ που αντικαθιστά τον κύριο Καντέρα Ρίφ, τον κύριο Ζων Ζακόμπ Μπισέπ που αντικαθιστά τον κύριο Πασκάλ Κανφά και τον κύριο Κάριμ Ζεριμπή που αντικαθιστά τον κύριο Βανσάν Πεγιόν. Καλωσορίζω τους νέους συναδέλφους και υπενθυμίζω στους κυρίους Ανδρίου Μπισέ και Σεριμπή ότι συμμετέχουν στα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνεδριάσεις του στο βαθμό, με πλήρη άσκηση δικαιωμάτων, στο βαθμό που ε, δεν υπάρχει ασυμβατότητα ως προς την άσκηση του λειτουργήματος αυτού. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Ο κύριος Σεριμπή επίσης μου ανακοίνωσε ότι έχει προσχωρήσει στην ομάδα των Πρασίνων. Οι αρμόδιες αρχές